good morning. And I'm just going to do the announcements while you get settled down. Καλημέρα, καθίστε παρακαλώ. Να μιλήσουμε για το γλωσσικό, μαλτέζικα, κροατικά και γκέλικ δεν θα έχουμε σήμερα. Και όσον αφορά την έγκριση των συστάσεων των συντονιστών, έχουμε κάποια πράγματα για τη Λίμπε, έτσι, Φανάρς ΕΛΚ. γίνεται εισηγητή για τη διαλειτουργικότητα, Νάτζια Ποτάλκ, για την έκθεση δίας πρωτοβουλία για τι ελάχιστε ε, προεγραφές για τι ε, μειονότητε. και ο κύριος ε, Νάγκη ορίστηκε εισηγητή για το δεύτερο τμήμα της διαλειτουργικότητας Στις 10.30 ψηφίζουμε, να ξέρετε. Εντάξει, να έχετε τις κάρτες σας παρακαλώ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ χαίρομαι που μπορώ εδώ να καλωσορίσω τους δύο συνεισηγητές μου, την κυρία, μάλλον τους δύο συμπροέδρους μου, την κυρία Μακάβεν και τον κύριο Μακάλιστερ, για τη συζήτηση που θα έχουμε εδώ όσον αφορά τις εξελίξεις για ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Ασφαλή Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση. Έχουμε εδώ την προσκεκλημένη μας, την Διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού για την Μετανάστευση, την κυρία Μισελ Κλάιν Σόλομον. Ευχαριστούμε που ήρθατε για τη συζήτηση αυτή που θα κάνουμε μεταξύ μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση αυτή για το Παγκόσμιο Σύμφωνο έχει Ω εξή, καταρχήν να σα πω πώ θα διεξαχθεί σήμερα η συζήτησή μα. Έχουμε εκπροσώπου από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, από την ε, Βουλγαρική Προεδρία που μπορούν να πάρουν το λόγο, από την Πρεσβεία του Μεξικού επίση έχουμε εδώ πέρα εκπροσώπου. Γιατί είναι και αυτοί αυτό που λέμε διαμεσολαβητές όσον αφορά το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Και για το παρακολουθείτε αυτό το θέμα πρόκειται για την συνέχεια που δίνεται στη δήλωση της Νέας ε, ε, Υόρκης που εγκρίθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου του 2016. Και είναι δύο, μία για τους πρόσφυγες και μία για τους μετανάστες. Και οι τρεις επιτροπές μας δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την υπόθεση του Παγκοσμίου Συμφώνου με διάφορες συναντήσεις μας που έχουν αφιερωθεί σε αυτό το θέμα, ακριβώς επειδή έχει μεγάλη σημασία όλο το ζήτημα της μετανάστευσης και στη συζήτηση θα φανεί γιατί. Και ποιος μπορεί να μας τα πει καλύτερα από την προσκεκλημένη μας, την Γενική Διευθύντρια του Παγκοσμίου Συμφώνου για την Ασφαλή Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Η Μισελ λοιπόν το 19 Σεπτεμβρίου 2016 μίλησε στον ΟΗΟ όσον αφορά το παγκόσμιο αυτό σύμφωνο για την ασφαλή ομαλή και τακτική μετανάστευση. Γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της μετανάστευσης. Πριν δώσω το λόγο στη Μισελ, Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μακάλιστερ, ώστε και εκείνος ε, να κάνει μια μικρή εισαγωγή. Μετά θα έχουμε την κυρία Μακάβεν από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Κλοντ Μωράες. Καλημέρα σε όλους τους συναδέρφους. Χαίρομαι για την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται να έχουμε μια συζήτηση από κοινού των τριών επιτροπών μας όσον αφορά το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο βέβαια δεν αφορά μία μόνο κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά είναι σημαντικό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον όσον αφορά το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, είναι σωστό χώρο να συζητηθεί αυτό, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη τοποθέτηση εν ώψη των διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί αυτή τη διαδικασία από κοντά. Ήδη από το 2016 με την Σύνοδο του ΟΙΕ για αυτό το θέμα και τις δραστηριότητες απολογισμού. Οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν στα τέλη αυτή της χρονιάς. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε το θέμα αυτό του Παγκόσμιου Συμφώνου με την κυρία Σόλομον. Οπότε θα δώσω το λόγο στην ε, προσκεκλημένη μας, αν συμφωνείς και εσύ Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο και τους τρεις πρόεδρους. Πράγματι είναι τιμή για μένα που μπορώ και βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές για την πρόσκλησή σας να έρθω σε αυτήν την κοινή σας συνάντηση. Είναι μια ενδιαφέρουσα συγκυρία και σε διεθνές επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την μετανάστευση. Ο Βίλιαμ Σίγκλεν θα ήθελε πάρα πολύ να έρθει επίσης εδώ και να σας μιλήσει, ζητά συγγνώμη όμως που δεν μπόρεσε. Υπάρχουν λοιπόν τεράστιες ροές μεταναστών και προσφύγων που έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια τόσο στη Μεσόγειο όσο και αλλού και θέτουν το ζήτημα το κατά πόσο έχουμε κατάλληλες εθνικές αλλά μάλλον εθνικά και διεθνή συστήματα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κινητικότητα. Οπότε έφτασε η στιγμή όλοι να εξετάσουμε την στάση μας, να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται σε τοπικό, σε εθνικό, σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Και όπως λέμε, στα πλαίσια ε, της συνέλευσης του ΟΗΕ προκειμένου να υπάρξει ένα παγκόσμιο σύμφωνο για την ασφαλή ομαλή και τακτική μετανάστευση. Κατά την άποψη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, το σύμφωνο αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στους ηγέτες μας Όντω να πάρουν τι σωστέ αποφάσει και να έχουν μια ισορροπημένη προσέγγιση απέναντι στη μεταναστευτική πολιτική. Και να μην σκέφτονται μόνο τι θα γίνει βραχυπρόθεσμα, να μην σκέφτονται μόνο τι εκλογέ, αλλά να σκέφτονται και το μακροχρόνιο συμφέρον, το τι συμφέρει να πάνω σαν απόφαση μακροπρόθεσμα. Σίγουρα και το κοινοβούλιο σα έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Αλλά όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται να νιώσουν ότι προστατεύεται η πολιτισμική τους ταυτότητα και η ταυτότητά τους γενικά. Και όλα αυτά τα εξετάζει το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Θέλω να υποφελθώ λοιπόν από αυτή την ευκαιρία για να σας παρουσιάσω τα θέματα τα οποία μας απασχολούν γενικότερα και να σας δώσω μια προοπτική για το μακροπρόθεσμο επίπεδο. Πρώτα απ' όλα, ποιε είναι οι προκλήσει κλειδί που αντιμετωπίζουμε ω διεθνή κοινότητα. Δεύτερον, τι προσπάθειε ε, πρέπει να γίνουν για το παγκόσμιο αυτό σύμφωνο. Και το τρίτο, ποιο είναι ο ρόλο των βουλευτών για να προωθήσουν πολιτικέ που είναι πιο δίκαιε, πιο έξυπνε, πιο ανθρώπινε για να αντιμετωπιστεί το μεταναστευτικό. Πρώτα λοιπόν για τι προκλήσει. Τρει θα λέγω ότι είναι. Και η πρώτη είναι η δημογραφική πρόκληση. Και εδώ οι δημογραφικές αλλαγές έχουν τεράστιες επιπτώσεις στις οικονομίες μας, στις κοινωνίες μας, όχι μόνο σήμερα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Και αυτό το βλέπουμε σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως στην Ευρώπη, όπου υπάρχει δημογραφικό ζήτημα. Γι' αυτό ίσως πρέπει να πάμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σε πολλές αφρικανικές χώρες ο μισός πληθυσμός είναι κάτω των 25 και προβλέπεται ότι το 25% του πληθυσμού θα βρίσκεται στην Αφρική το 2050. Οπότε αυτή η δυναμική θα οδηγήσει σε δύσκολες πολιτικές επιλογές. Σίγουρα η μετανάστευση ποτέ δεν θα αποτελέσει την μόνη λύση στην δημογραφική συρρήκνωση που αντιμετωπίζουν κάποιες χώρες ή περιοχές, αλλά σίγουρα και η μετανάστευση αποτελεί μέρος της λύσης. Δεύτερον, η μετανάστευση θα συνεχίσει να επηρεάζει τις κοινωνίες μας και τη σύνθεσή τους. Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να τα βρούνε, να το δεχτούν και να αντιμετωπίσουν τη θρησκευτική και άλλες διαφοροποίησεις. Βέβαια, όταν υπάρχουν τοξικά αφηγήματα όσον αφορά την μετανάστευση, αυτό οδηγεί σε αρνητικές συνέπειες. Ξανά και ξανά έχει φανεί ότι τελικά οι μετανάστες οδηγούνται σε χαμηλότερη εγκληματικότητα από ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί στις χώρες μας. Αντίθετα, βοηθούν με δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και αυτή είναι η λύση. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε ο δημόσιος λόγος να είναι πιο ισορροπημένος και να είμαστε πιο αντικειμενικοί όταν μιλάμε ως πολιτικοί. Και όσον αφορά την ποικιλομορφία, θα πρέπει πρέπει να προωθήσουμε την ε, μετανάστευση, αλλά από μόνη της δεν θα αντιμετωπιστεί η ποικιλομορφία σωστά. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες στα σχολεία, στα κοινωτικά κέντρα, στις οικογένειες. Τώρα η δεύτερη πρόκληση που συχνά βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης είναι οι καταστροφές ε, λόγω των οποίων μετακινείται ο κόσμος. Και όντως, δυστυχώς, τέτοιες αιτίε είναι όλο και περισσότερες τα τελευταία χρόνια. Αλλά σε σχέση με τη μετακίνηση του πληθυσμού, λιγότερο από όσο θα φανταζόταν κανείς. Οι ε, οικονομικές και γνώσεις υποθέσεις του Ιαϊπαν μίλησαν για 288.000 μετανάστες σήμερα. 20 εκατομμύρια όμως είναι οι πρόσφυγες. Και υπάρχουν και 40 εκατομμύρια που μετατοπίζονται στο εσωτερικό των ίδιων των χωρών τους. Το αποτέλεσμα με αυτές τις μικτές ροές μεταναστών προσφύγων και μεγάλες ε, ε, ροές Γίνονται μετακινήσεις, χωρίζονται οικογένειες, μένουν παιδιά ασυνόδευτα. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε πολιτικές που να αναγνωρίζουν τους μεγάλους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όλοι κατά τις διαδρομές τους και να λάβουμε υπόψη μας την εκμετάλλευση που υφίστανται συχνά και ότι πολλοί από αυτούς πληρώνουν την ίδια τη ζωή τους. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο λοιπόν να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που μετακινούνται και να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους. Η εμπειρία δείχνει ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα δεν φτάνουν. Η διεθνής κοινότητα θα είναι πιο αποτελεσματική αν λάβει υπόψη της τη μετανάστευση πιο μακροπρόθεσμα, με μακροπρόθεσμες πολιτικές όσον αφορά την κινητικότητα. Να λάβει υπόψη τις αιτίες που οδηγούν στη μετανάστευση. Ακόμα και ε, τις, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και βέβαια τις συνέπειες ε, μιας ε, καταναγκαστικής μετανάστευσης τελικά. Και πρέπει να βρεθούν νόμιμοι οδοί μετανάστευσης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας με υποχρεώσεις για προστασία. Τότε θα υπάρχουν λιγότεροι κίνδυνοι και θα προστατεύονται καλύτερα τα ευάλωτα άτομα γιατί θα ακολουθούν τις νόμιες οδούς. Τώρα θα επανέλθω στο Παγκόσμιο Σύμφωνο και αυτό είναι το καλό νέο. Το Σεπτέμβριο πέρυσι τα Ηνωμένα Έθνη είχαν την πρώτη τους διάσκεψη για να συζητήσουν το θέμα των μεγάλων αυτών μεταναστευτικών ε, ε, ροών και κατέληξε σε μία δήλωση που αναγνωρίστηκε από όλες τις χώρες μέλη ως μία ανάγκη για συνολική προσέγγιση και επιτρέπει να δημιουργηθούν δύο παγκόσμια σύμφωνα. Το ένα για τους ε, μετανάστες και το άλλο για την ασφαλή ομαλή και τακτική μετανάστευση. Μάλλον το πρώτο για τους πρόσφυγες και το δεύτερο για την ομαλή και τακτική μετανάστευση. Ήδη είχαμε τα πρώτα δείγματα από τον ΟΗΕ αυτές τις μέρες και όπως είπε και ο Πρόεδρος εδώ, το Παγκόσμιο αυτό σύμφωνο αφορά μια διαδικασία. Τη Δευτέρα οι διαμεσολαβητές, το Μεξικό και η Ελβετία δηλαδή, θα μας παρουσιάσουν το λεγόμενο Zero Draft. Και μετά θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις κάθε μήνα από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο στη Γενέβη. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο λοιπόν πιστεύω ότι είναι μια πολύτιμη ευκαιρία για τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να αφοσιωθεί σε αυτό το κοινό όραμα που είναι να αντιμετωπιστεί η μετανάστευση, να γίνεται σε θελοντική βάση και όχι κάτω από απελπισία και οι κυβερνήσεις να έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τη μετανάστευση με τρόπο επωφελή τόσο για τους μετανάστες όσο και για τις χώρες φιλοξενίας και χρειάζεται συνεργασία βέβαια και με τις χώρες πρόλευσης. Και έρχομαι στο τρίτο μου στοιχείο που είναι ο ρόλος των βουλευτών και τι εσείς μπορείτε να κάνετε για όλα αυτά. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι βουλευτές έχουν ισχυρή φωνή και πρέπει να έχουν ισχυρή φωνή τόσο στην ε, ε, εκπόνηση όσο και στην εφαρμογή του Παγκοσμίου αυτού Συμφώνου για την μετανάστευση. Και αυτό το οποίο έχω να σας ζητήσω είναι με σοφία να χρησιμοποιήσετε τις εξουσίες που διαθέτετε. Πρώτον, εκπόνηση πολιτικής να χρησιμοποιήσετε λοιπόν την ε, πολιτική σας, την εφαρμογή της, αλλά και ε, τα κονδύλια που μπορείτε να διαθέσετε. Ο μετανάστης θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο και διαχείριση της μετανάστευσης και οι μετανάστες να λαμβάνονται υπόψη στα εθνικά σχέδια στρατηγικής, σε σχέδια για την στέγαση, σε σχέδια για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, αλλά και σε κοινωνικές, όπως είναι πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία. Ζητούμε από τους βουλευτές, εθνικούς και ευρωβουλευτές, να υπάρξει ε, ένα καθεστώς ε, θεωρήσεων, όπως ζητάει ο οργανισμός μας, για τους ευάλωτους μετανάστες, για αυτούς που χρειάζονται ειδική προστασία και να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις χώρες ε, μέλη βάσει των όσων ισχύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μπορούν αυτό να το κάνουν με ασφαλή τρόπο. Οι βουλευτές επίσης μπορούν να βοηθήσουν σε μια νέα προσέγγιση των χωρών μελών πολλά διαφορετικά υπουργεία και αρχές είναι αρμόδιες για θέματα που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει κατακαιρματισμός αλλά συνεργασία. Πρέπει η μετανάστευση να συμπεριληφθεί επίσης τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2030. Υπάρχει δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ανάπτυξη και την ε, στρατηγική της Ευρώπης για την ασφάλεια. Τώρα το άλλο που μπορεί να κάνετε είναι ότι μπορείτε να αλλάξετε τα τοξικά αφηγήματα που υπάρχουν για τη μετανάστευση. Να φροντίσετε να είναι πιο ισορροπημένα αυτά τα οποία ακούγονται. Δυστυχώς ο κόσμος πολύ συχνά ακούει ανεύθυνη ρητορική ορισμένων πολιτικών και αποδέχεται την αρνητική εικόνα. Οπότε οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να υπενθυμίσουν στους πολίτες τους πώς έχει συνεισφέρει η μετανάστευση στην οικονομική και κοινωνική διάσταση, αλλά και ότι πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις προς όφελος και των ε, ε, μεταναστών και των κοινοτήτων που τους ε, φιλοξενούν. Οι πόροι τώρα. Οι πόροι μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση στο μεταναστευτικό και θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Πρώτον, ένταξη και κοινωνική πολιτική όπως είπα και πριν, απαιτεί επενδύσεις προκειμένου να αποδεχτούμε τους μετανάστες. Πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, κυρίως στην υγεία, την εκπαίδευση και την ε, κοινωνική αρρωγή. Ε, Όλοι γνωρίζουμε ότι πάντα θα υπάρχουν περισσότεροι που θέλουν ε, να έρθουν στις χώρες μας από ό,τι μπορούν να επιτρέψουν οι κυβερνήσεις. Ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες και βάσει αυτών κάποιοι θα πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες τους. Είναι βασικό στοιχείο και αυτό της μεταναστευτικής πολιτικής. Όσο γίνεται περισσότερο βέβαια, οι επιστροφές αυτές θα πρέπει να είναι σε θελοντική βάση και να προσφέρεται κάποια βοήθεια σε αυτούς, κάποιο ποσό, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν ε, πιο εύκολα στις τοπικές τους κοινότητες, να παραμείνουν στις χώρες δηλαδή όπου έχουν επιστρέψει. Οι διαβουλεύσεις πάντως για το ετήσιο πλαίσιο προσφέρουν μια ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει σε δράση τις επιθυμίες της με τα κατάλληλα οικονομικά μέσα και έτσι να πετύχουν οι φιλοδοξίες σας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συνεισφέρει ως αρμόδια αρχή επί του προϋπολογισμού για να υλοποιηθεί αυτό. Και θα ολοκληρώσω κυρίες και κύριοι με κάποιες σκέψεις. Η μετανάστευση ήρθε για να μείνει. Αντί λοιπόν να τη βλέπουμε σαν ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε, καλά θα κάνουμε να τη δούμε σε μια πραγματικότητα ανθρώπινη που πρέπει να διαχειριστούμε. Μετά την έκθεση του Γενικού Γραμματέα που μιλάει για τη μετανάστευση για όλους, πρέπει να ξέρουμε ότι η μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για όλους μας και να αναγνωριστεί ότι η ανθρώπινη κινητικότητα αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της ανθρωπότητας της προηγούμενης, της ιστορικής και της μελλοντικής. Συμφωνούμε λοιπόν και εμεί, ο οργανισμός μας, με τον ε, Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και βάσει αυτού θα παρακολουθήσουμε το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Όσο προχωράει η διαδικασία στι διαπραγματεύσεις, σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε συνεργασία μεταξύ μας και κοινή δράση για να αναπτύξουμε μια πραγματικά κοινή τοποθέτηση και στάση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη θα πρέπει να ηγηθούν στις διαπραγματεύσεις αυτές και να διασφαλίσουν ότι θα εγκριθεί μια φιλόδοξη συμφωνία με ένα ενιαίο πλαίσιο με κοινέ αρχές, δεσμεύσει και κατανόηση μεταξύ των χωρών μελών και αυτό για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση και κυρίως με τους στόχους της βιωσιμότητας στο σημείο 17 που μιλάει για ασφαλή, ομαλή, τακτική και υπεύθυνη μετανάστευση. Άρα χρειαζόμαστε υπεύθυνε πολιτικές μετανάστευσης τις οποίες θα διαχειριζόμαστε και καλά. Χαιρόμαστε λοιπόν που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για αυτά. Θα υπάρξει και νέα συνάντηση για να επεκταθούμε περισσότερο σε αυτά τα ζητήματα όταν θα έχουμε το σχέδιο Zero. Και χαιρόμαστε πολύ που εσείς οι Ευρωβουλευτές μπορείτε να αναλάβετε ηγετικό ρόλο σε αυτήν την ιστορική σημασία διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κυρία Σας ε, Ευχαριστούμε που αναφερθήκατε στο ρόλο των βουλευτών και στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Θέλω να θυμίσω μόνο ότι και οι τρεις συναρμόδιες επιτροπές ε, από την 16η Σύνοδο για τους μετανάστες και τις πρόσφυγες έχει εμπλακεί ενεργά στη διαδικασία και σε σχέση με την παγκόσμια δήλωση και φυσικά θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεκης τις διεθνείς ε, διαπραγματεύσεις και συνομιλίες που θα αρχίσουν ε, στα τέλη του Φεβρουαρίου μετά από την δημοσίευση του αρχικού σχεδίου του Zero Draft σε λίγες μέρες. Πριν αρχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση για τα μέλη και των τριών επιτροπών, ναι, δηλώστε συμμετοχή. Θα ακούσουμε σύντομα κάποιον από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και από τη Βουλγαρική Προεδρία. Παρακαλώ να είστε σύντομοι όμως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάρα πάρα πολύ σύντομος θα είμαι. Ε, Δύο-τρία σημαντικά σημεία θέλω να επισημάνω γιατί δραστηριοποιούμαστε σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη όλους ιδιαίτερα σε αυτούς τους τομείς. Μετά την δήλωση της Νέας Υόρκης το 2016 ε, διαπιστώνουμε με ικανοποίηση πως τα κράτη-μέλη υιοθετούν μια κοινή προσέγγιση και αντίδραση ως προς αυτή την ε, ε, ομολογουμένως ευπρόσδεκτη δήλωση σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και κυρίως με, την με τις εκπεριτροπείς προεδρίες στις διάφορες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, ε, το, κυρίως με την υψηλή ομάδα σύλλου και μετανάστευσης. Κάνουμε μία ε, απογραφή σε σχέση με όλα όσα έχουμε και που συνιστούν την κοινή συνεννόηση ε, μεταξύ κρατών μελών. Όχι ότι ε, οδηγούμαστε προς ε, κοινέ κατευθυντήριες γραμμές, απλώς έχουμε μία σειρά από κοινά σημεία για τα οποία τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει ότι θα συνεργαστούν για να μεγιστοποιήσουμε τη διαφάνεια ως προς την προεργασία που γίνεται για τις διαπραγματεύσεις και για να εξασφαλίσουμε ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις μας κυρίως προς τους ε, στόχους της χιλιετίας ε, και για τις εσωτερικές προκλήσεις αλλά και την εξωτερική διάσταση ε, της πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης. Δεν θα υπησέλθω τώρα σε λεπτομέρειες για το τι κάνουμε, διότι δεν χρειάζεται εγώ να παρουσιάσω τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις των δύο κρατών μελών, απλώς ε, μπορεί να μιλήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα αναφερθώ στην εξωτερική διάσταση. Ε, έχουμε δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερε επαφές μας με τις τρίτες χώρες και θέλω εντάχει να αναφερθώ στη, ε, τα αποτελέσματα του Αμπιτζάν για την ε, κατάσταση στην ε, Λιβύη, στην Σύνοδο Αφρικανικής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΗΕ και Έχουμε την δέσμευση των Αφρικανικών χωρών και την πρόοδο που έχουν σημειώσει ως προς την υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης, δηλαδή έχουν επιληφθεί το ζητήμα όπως το ζητήσαμε, και υποστηρίζουν το, τη δουλειά του IOM, τη, του, διεθνής, Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσης. Ε, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ, με την ε, Οικογένεια Αφρικανικών Χωρών, με την Αφρικανική Ένωση και με τα κράτη-μέλη, έχουμε μια κοινή δυναμική που θα μας οδηγήσει στην ε, διαμόρφωση του Παγκοσμίου Συμφώνου. Πιστεύω ότι ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση και εκφεύγουμε λίγο από το, το, κλασικό φύγημα και προσπαθούμε να με ρητσικέλευτο τρόπο να σημειώσουμε πρόοδο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε τώρα ε, συντομία και την ε, Βουλγαρική Προεδρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητά μέλη των τριών επιτροπών, αγαπητοί συναδέλφοι, να σας ενημερώσω ε, τι, για τα πορίσματα του Ατύπου Συμβουλίου Δικαιοσύνης Εσωτερικών Υποθέσεων για το Παγκόσμιο Σύμφωνο Μετανάστευσης στις 25 Ιανουαρίου στη Σόφια. Ε, ενεγράφει στην ημερήσια διάταξη του Ατύπου Συμβουλίου, διότι η κυρία για η ειδική εκπρόσωπος του ΕΕ για την διεθνή μετανάστευση, μετήχε στο Ατύπου Συμβούλιο και κατά την προετοιμασία του Συμβουλίου, η κυρία Άρμπορ συμμετείχε στην συζήτηση που έγινε από του υπουργού Εσωτερικών και τους υπουργού Αρμοδίους για θέματα μετανάστευση. Ε, και όλοι συμφώνησαν ότι είναι αμοιβέω επωφελή η διαδικασία διότι έτσι γνωρίζουν οι υπουργοί τα απορίσματα των εργασιών του ΙΕ για το μελλοντικό παγκόσμιο σύμφωνο και ταυτόχρονα ε, κατεγράφησαν ε, πολύ σημαντικά στοιχεία προόδου ε, που θα ανακύψουν και στις επικείμενες διαπραγματεύσεις. Δυστυχώς όμως, τελευταία στιγμή η κυρία Άρμπορ δεν μπόρεσε να έρθει. Παρόλα αυτά, ε, οι επόλοιποι προσκεκλημένοι ήρθαν, αναπληρωτής διευθυντής ε, η κυρία Λόρα Τόμσον από τον IOM, ε, ο αναπληρωτής με κύριος Τιούρκ, ύπατος εκπρόσωπος για τα θέματα μετανάστευσης και ε, για να ευθυγραμμίσουμε τη συζήτηση σε σχέση με τους στόχους μας παρουσιάσαμε εμείς ένα έγγραφο με τρεις ερωτήσεις για το περιεχόμενο, για την ισορροπία ανάμεσα στους στόχους και για την εφαρμογή του GCM. Ήταν πολύ ζωηρή η συζήτηση, έγιναν ε, αρχικές τοποθετήσεις ε, των προσκεκλημένων μας ε, που ε, έθεσαν και τις βασικές κατευθυντήρες αρχές του μελλοντικού συμφώνου, δηλαδή συγκεκριμένα να υπάρχει ισορροπία, να υπάρχει η προσέγγιση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο κεντρικός ρόλος της δήλωση, της, της Νέα Υόρκης, ο ρόλος της διεθνούς συνεργασίας και η ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στις αρχές της δήλωσης Νέας Υόρκης του Παγκοσμίου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και για τον Διεθνό κοινών πολιτικών στον τομέα της μετανάστευσης. Τονίστηκε πόσο σημαντικό παίκτη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα και έχει ήδη συνεργαστεί επικοδομητικά στην ε, προπαρασκευαστική φάση. Ε, η συζήτηση οδήγησε σε κοινή σε συνένεση και συνεννόηση σε σχέση με αυτές τις βασικές ε, κατευθυντήριες αρχές που προανέφερα. Η προσθέμενη αξία για καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών του Παγκοσμίου Συμφώνου, το στοιχείο ότι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές όλων των κρατών μελών και πρέπει να βασίζεται σε μια κοινή προσέγγιση προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ιδιαίτερη εστίαση σε ευπαθείς ομάδες, ανάγκη διαφοροποίησης φυσικά ανάμεσα στις δύο κατηγορίες προσφύγων και μεταναστών. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο πρέπει να τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες μετανάστευσης για να έχουμε τα ε, προσφορότερα μέτρα για την τακτική μετανάστευση και την αντιμετώπιση της εμπορίας ε, ανθρώπων και ε, της ε, δράσης των διακινητών ασφαλής οδή μετανάστευση σε βάση των διεθνών αρμιδιοτήτων για τη συνεργασία των κρατών μελών για την επανεισδοχή των υπηκόων τους. Επίσης, θα κοινωνική συμπερίληψη των μεταναστών στις χώρες επιδοχής Οι Υπουργοί Εσωτερικών επανέλαβαν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή και υπεύθυνη διεθνή συνεργασία για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των ε, ηλμένων δεσμεύσεων. Και επίση συμφωνία σε σχέση με το ότι πρέπει να, έχει, να μιλάει με μια φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την προπαρασκευαστική βάση των διαπραγματεύσεων. Ε, στη... Θα σας παρουσιάσουμε τα απορίσματα των συζητήσεων σωμάτων εργασίας ε, του Συμβουλίου Ε, για τις, για τις επικίνδυνες διαπραγματεύσεις ε, στη Νέα Υόρκη. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στο να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Σας ευχαριστούμε. Ας περάσουμε τώρα στα μέλη των Επιτροπών. Παρακαλώ από τις τρεις Επιτροπές, ΑΦΕΝΤΕΒΕ ε, και ΛΥΒΕ, δηλώστε ποιοι θέλετε να συμμετάσχετε. Α, η κυρία Μέτσολα έφυγε. Ωραία, αρχίζουμε. Όχι, εδώ είναι τα λέει. Τα λέει με, ένα, με κάποιον άλλον από τη ΛΥΜΠΕ. και οι άλλοι δεν συζητάνε και η ΣΥΠΟΛ πάει και αυτή. Α, Σαρτζεντίνη. Ε, και να διαφυλάξετε τη φήμη της Λίμπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν ήξερα ότι είμαι και δεύτερη στον κατάλογο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την κυρία Κλάιν Σόλομιν, γιατί νομίζω ότι διαπιστώνεται αυτή τη σχιζοφρενική κατάσταση που βιώνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα τελευταία λόγια τη εκπροσώπου του Συμβουλίου τη Βουλγαρική Προεδρία ήταν ότι συνεχίζουμε να μιλούμε με μία φωνή. Ε, προσωπικά φρονώ ότι μιλούμε ίσως με μία φωνή στη Νέα Υόρκη, αλλά με άλλη φωνή όταν ε, ε, συζητούμε στα Συμβούλια Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και υπάρχει συζήτηση μεταξύ Υπουργών Εσωτερικών. Η... Όλη η συζήτηση για το Παγκόσμιο Σύμφωνο ε, εξωτερικά φαίνεται ότι καλύπτει όλα τα βασικά στοιχεία, δηλαδή ότι κατανοούμε ότι η Ευρώπη είναι μια ήπειρος μετανάστευσης, ότι οι νόμιμες μεσοδοί βοηθούν αυτούς που πραγματικά θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας και πρέπει να παρέχουμε νόμιμους διάβλους. Αλλά οι πολιτικές που εφαρμόζουμε σε εσωτερικό επίπεδο δεν αντιχούν αυτή τη συνεννόηση, αυτή την αντίληψη. Και νομίζω ότι το εξή θα έπρεπε να πούμε στη Βουλγαρική Προεδρία. Πώ μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε την αντίληψη που έχουμε για τη μετανάστευση ω παγκόσμιο φαινόμενο και εμεί θα πρέπει να συμμετέχουμε ω Ευρώπη και με τι πολιτικέ που έχουμε αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, η όλη διαδικασία επαναγκατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει συνεννόηση με τα κράτη-μέλη και να λέμε ότι δεν μπορούμε να μιλούμε μόνο για το μέγιστο αριθμό των ατόμων που δικαιούνται επαναγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν είναι κάποιο να διατεθειμένος να συζητήσει και τον ελάχιστο αριθμό ανθρώπων που αναζητούν έναν ασφαλή χώρο εδώ στην Ευρώπη. Και επίσης θα ήθελα να καταλάβω κατά πόσον η κυρία Κλάιν Τσόλομον αναφέρεται σε ευρωπαϊκό ε, ευρωπαϊκή θεώρηση διαβατηρίων για ανθρώπους που είναι ευάλωτοι και όχι μόνο για αυτούς που κάνουν αίτηση για καθεστώς ασύλου. Πώς το βλέπετε εσείς, διότι αυτή τη στιγμή ούτως έλος δίνουμε μάχη για να αντιληφθούν τα κράτη-μέλη ότι χρειάζονται χώρο, χρειάζονται θέση και οι πρόσφυγες. Πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε αυτά όταν υπάρχουν δύο διαφορετικά σύμφωνα και να μην έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ μεταναστών και προσφύγων. Ευχαριστώ, Τζούντιθ. Συνάδελφοι, δύο λεπτά το πολύ ο καθένας γιατί είναι μακρύς ο κατάλογος και πρέπει δέκα και μισή να έχουμε τελειώσει γιατί έχουμε ψηφοφορία. Η κυρία Λόχπίλτερ στη συνέχεια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την κυρία Κλάιν Σάλομον για την παρουσίαση που έκανε για τη δήλωση της Νέας Υόρκης. Ο στόχος είναι η προστασία και η ενίσχυση των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων. Και όπως είπατε, είναι γι' αυτό ιδιαίτερα σημαντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν εξετάζουμε αυτή την πολιτική βλέπουμε όμως ότι μονομερός εστιάζεται στην καταπολέμηση των παρανόμων μεταναστών και την αποτροπή των μεταναστευτικών ροών από τρίτε αντί να ενθαρρύνει την νόμιμη και την τακτική μετανάστευση. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Σε ποια μέσα θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε, ποιες δυνατότητες υπάρχουν για να αλλάξουμε την αιστεία στην κατεύθυνση αυτής της πολιτικής. Είπατε ότι θα πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μια τέτοια προσέγγιση όμως δύσκολο το βλέπω. Δεύτερη ερώτηση, ε, ο στόχος αυτού του Παγκοσμίου Συμφώνου Μετανάστευσης είναι να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη που υποδέχονται πάρα πολλούς πρόσφυγες μεγάλες μεταναστευτικές ροές. Όμως αυτό έχει και ως επίπτωση ότι ε, μένουν σε κέντρα υποδοχής ε, για πάρα πολύ καιρό οι μετανάστες. Για το 2016 πάνω από 5 εκατομμύρια μετανάστες ε, μένουν πάνω από 10 χρόνια σε κέντρα υποδοχής χωρίς καμία δυνατότητα να αποκτήσουν την ηθαγένεια, χωρίς καμία μελλοντική προοπτική. Πώς το αξιολογείτε εσείς και πώς μπορείτε να το συνδυάζετε αυτό με την δήλωση της Νέας Υόρκης. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και βεβαίως να ευχαριστήσω και την κυρία Κλάιν Σόλομον για την παρουσίαση που μας έκανε για την πρόοδο σε αυτή την πολύ σημαντική διαδικασία. Ήμουνα με κάποιους άλλους συναδέλφους στη Νέα Υόρκη για την πρώτη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για τις μεγάλες μετακινήσεις ε, των ε, μεταναστών και των προσφύγων και υπήρχε πολύ μεγάλο επίπεδο φιλοδοξίας. Αλλά οι αλλαγές στη γεωπολιτική κατάσταση νομίζω ότι θέτουν αυτές ε, τις φιλόδοξες ε, προτάσεις σε κίνδυνο και είδα και το θέμα της έγκρισης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και θα ήθελα να τα συνδυάσω και τα δύο. Ε, νομίζω ότι έχουν αντίκτυπο και στις δύο διαδικασίες με τρόπο που θα έπρεπε να μας ανησυχεί, με τρόπο που ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά να αναλάβει τα ενία και να πρωτοστατήσει στην εφαρμογή και την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και ε, την εφαρμογή αυτού του Παγκοσμίου Συμφώνου. Πρέπει όμως να πω ότι συμφωνώ με ε, τις ανησυχίες της συναδέλφου Αργεντίνη διότι δεν μιλούμε με μία φωνή. Και αν όντω μιλούμε με μία φωνή, ε, φοβάμαι για αυτά που λέμε. Φοβάμαι ότι δεν λέμε τα σωστά πράγματα. Και αν όντω θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο τη άρνηση, αρνούμαστε την πραγματικότητα, αρνούμαστε τα πραγματικά στοιχεία. Εσεί αναφερθήκατε σε μία προσέγγιση βάση αποδείξεων στη μετανάστευση. Θα το ήθελα πολύ να το δω αυτό, ακόμα και εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά πολύ συχνά δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Και αρνούμαστε και το γεγονό ότι η μετανάστευση ήρθε για να μείνει και ε, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλε πολιτικέ. Εάν δεν το δεχτούμε αυτό, δεν μπορούμε να είμαστε ε, αξιόπιστοι προ τα έξω. Δεν μπορούμε να αξιόπιστοι και στη Νέα Υόρκη όταν ζητάμε καλύτερο καταμερισμό ευθύνη ε, για τη μετανάστευση, αν δεν μπορούμε πρώτα να τα καταφέρουμε εδώ, στον οίκο μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καλό το γεγονός και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας ότι ε, ε, εμείς εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, και εν μέρη και στην Επιτροπή ΝΤΕΒΕ ασχολούμαστε με τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και τον Οκτώβριο καταφέραμε να εγκρίνουμε μια πολύ φιλόδοξη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου που θέτει προτεραιότητα για τα θέματα ασύλου στα διάφορα κράτη-μέλη. Και αυτό που προσπαθούμε να πούμε με αυτή τη μεγάλη πλειοψηφία είναι ότι είναι μια κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση που χρειάζεται κοινέ ευρωπαϊκές λύσεις. Είναι ένα καλό μήνυμα και ε, οι επιτροπέ αυτές θα αποτελέσουν σύμμαχό σα, όπως και το Κοινοβούλιο, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Κάτι τελευταίο και μια ερώτηση. Πώς επηρεάζει η αλλαγή κυβέρνησης ε, στις ΗΠΑ, Πολιτείες τις διαπραγματεύσεις. Θα υπάρχουν συνέπειες, θα δούμε και κάποιες άλλες χώρες ε, λόγω αυτού να φεύγουν από τη διαδικασία. Συνάδελφοι, παρακαλώ προσπαθήστε να τηρήσετε τα δύο λεπτά. Η κυρία Ζόφκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Δυστυχώς καθυστέρησα λίγο και δεν την άκουσα όλη, αλλά επειδή είμαι μέλο της ΔΕΒΕ και ταξιδεύω τακτικά ε, σε αυτές τις περιοχές, υπάρχει τεράστια εισρωή μεταναστών. Και θα ήθελα να σας θέσω μια ρεαλιστική ερώτηση. Ε, πριν από 20 χρόνια ήμουν και εγώ ε, πρόσφυγας ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγόμενη από την πρώην Ιουκοσλαβία. Και στις χώρες μας δυστυχώς υπάρχει πολύ μεγάλος λαϊκισμός. Πώς θα ανταποκριθούν τα Ηνωμένα Έθνη μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συντονίσουν την δημόσια διπλωματία και την βοήθεια βεβαίως, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής την αντιμετώπιση όλη αυτή τις κρίση, αλλά το ευρύ κοινό δεν αντιλαμβάνεται τι ακριβώς συμβαίνει και τι αντιμετωπίζουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ε, αναφέρεται στα Ηνωμένα Έθνη ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα της δημόσιας ε, διπλωματίας. Ε, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε στο κοινό τι ακριβώς κάνουμε και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις πηγές της μετανάστευσης με αποτυχημένα κράτη, αποτυχημένες χώρες και οι απαντήσεις που δίνουμε εδώ είναι ωραίες και ιδεολογικές και με μεγάλα ιδανικά, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Η Σιλβί Γκυγιόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση. Ε, συμφωνώ με πολλά από όσα ακούστηκαν, κυρίως από την Ellis Line ε, προλίγου και πάντα χαίρομαι να σας ακούω, να αναφέρεστε σε ένα φαινόμενο το οποίο είναι κυκλικό, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πηγή και τα αίτια της μετανάστευσης ε, και να μιλούμε και για την κοινή γνώμη και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και αποδέχονται κάποια πράγματα και είμαι και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη για όλα ε, αυτή την πολιτική για την ε, ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση. Πέραν των όσων ακούστηκαν ήδη, θα ήθελα να πω τα εξή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταφέρουμε να μιλήσουμε και για το θέμα της βίας ε, κατά των μεταναστών, των ετούντων άσυλο ή των προσφύγων. Ανεξάρτητα από το που βρίσκονται ή τι πορεία έχουν ακολουθήσει ε, τι μπορούμε να κάνουμε για τη μείωση αυτής της βίας ε, κατά αυτών των ανθρώπων και να αναφερθώ και σε τρεις διαστάσεις. Καταρχάς, ε, τι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ως εφαλτήριο για να μειώσουμε δραστικά τα περιστατικά βίας ε, κατά των μεταναστών που τον ετούν τον άσυλο ή των προσφύγων, ανεξάρτητα από τη φύση ή το που βρίσκονται ή το πώς ήρθαν. Τη δεύτερη ερώτηση που θα ήθελα να θέσω είναι η εξή. μήπως αυτό επηρεάζει και τα εν λόγω άτομα, αλλά η καταπολέμηση και της βίας ε, μπορεί να έχει και κάποιο αντίκτυπο και στην ίδια ε, τη χώρα και για τον, ε, την κοινή γνώμη και για αυτά τα οποία συζητήσαμε. Και όσον αφορά αυτούς που συμμετέχουν Μήπως ε, θα μπορούσε να είναι και ένας πολύ καλός άξονα κινητοποίηση να χρησιμοποιηθεί το θέμα αυτό και αυτοί οι οποίοι μας βοηθούν, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά ίσως και άλλοι ενδιαφερόμενοι, να μπορούσαν να βοηθήσουν για να μπορέσουμε πραγματικά να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πλήττονται από τη βία, αλλά και να αλλάξουμε και την ε, άποψη τη κοινή γνώμη. Ευχαριστώ. Η Κλέαρ Μουντι. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ελπίζω ότι εδώ πέρα φέρετε κλαυκά της Αθήνας. Δηλαδή είμαστε εμείς πεισμένοι για όλα αυτά που μας λέτε ήδη. Όντως υπάρχει το πρόβλημα της επικοινωνίας, πώς δηλαδή τις πολιτικές μας να τις εξηγήσουμε στις χώρες μας. Πάντως, αυτά τα οποία ε, με ενδιαφέρουν και που καλύψατε νωρίτερα, ένα από αυτά είναι το θέμα το δημογραφικό και το άλλο είναι το οικονομικό για να στηρίξουμε τη μετανάστευση στις χώρες μας. Αν δείτε τα στοιχεία για τα συνταξιδιωτικά ταμεία στις χώρες μας, το δείχνουν ξεκάθαρα γιατί οι περισσότερες χώρες χρειάζονται νέους να μπουν στην αγορά εργασίας τους, στις οικονομίες τους, γιατί δημιουργείται άλλη καταστροφή εκεί. εκεί που δεν τα καταφέρουμε είναι να στείλουμε το σωστό μήνυμα που θα αγγίξει τις καρδιές του κόσμου. Να εξηγήσουμε δηλαδή γιατί είναι σημαντικό και γιατί πρέπει μάλλον να αγκαλιάσουμε τη μετανάστευση αντί να την κατατροπώνουμε. Και αυτό βέβαια συνδέεται πολλές φορές με την ασφάλεια. Αυτό δηλαδή που ζητάω από σας πιο πολύ είναι να μας δώσετε βέλτιστες πρακτικές. Τι αναφέρεται στην ε, ανακοίνωση όσον αφορά τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για να μεταφέρουμε αυτά τα μηνύματα που θέλουμε πραγματικά να μεταφέρουμε. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Θέλω να συμφωνήσω με πολλούς συναδέρφους, λέγεται Μετσόλα, για το εξή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ψώσει τη φωνή του πολλές φορές και έχει επιμείνει για το ότι πρέπει να αναλάβουμε τα κατάλληλα βήματα προς τα μπρος. Είναι μια εντολή. Περάσαμε από μια σταθερή κατάσταση σε μια κατάσταση κρίσης. Τώρα σταθεροποιείται πάλι λαμβάνοντας υπόψη μας τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Όμως, όσον αφορά την ε, νόμιμη μετανάστευση, σε μια κατάσταση όπου δεν έχουμε καθημερινή κρίση με εκατοντάδες χιλιάδες να μας φτάνουν, θα έπρεπε να κοιτάξουμε να βρούμε μέτρα τα οποία να επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια αξιόπιστη πολιτική. Και συμφωνώ με την κυρία Σαρτζετίνη, όταν συγκρίνουμε το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο, ε, είμαστε πολύ μακριά από τον άλλον. Εμείς εδώ αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να προσφέρεται προστασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθείαν στους ανθρώπους αυτούς τους πιο ευάλωτους για να μην κινδυνεύουν ε, τη ζωή τους και να μην πνίγονται στις θάλασσές μας. Για να το κάνουμε όμως αυτό πρέπει να δούμε τις χώρες μέλη που έχουν μια καλή παράδοση προστασίας χιλιάδων ανθρώπων που βρίσκονται στα εδάφη τους, είτε επειδή είναι ευάλωτοι, είτε επειδή θέλουν να καλύψουν τις, ε, τα οικονομικά τους κενά, τα δημογραφικά κλπ. Πρέπει να το δούμε αυτό σαν μια πιθανή λύση. Σε κάποιες χώρες γίνεται κατανοϊκό, αλλού δεν γίνεται κατανοϊκό, γιατί δεν έχουν παράδοση σε τέτοια γιατί έχουν ήδη εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπους ε, που χρειάζονται προστασία στο εδαφο του. Πάντως, ή που θα είμαστε σοβαροί για να εντοπίσουμε τις τρίτες χώρες από όπου ε, μπορούν να έρθουν άνθρωποι και να χαίρουν προστασία από εμά βάσει τη συνθήκη τη Γενέβης, αλλιώ δεν θα καταλήξουμε πουθενά και που θα ολοκληρωθεί άλλη μια θητεία τότε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την οποία θα λέμε αργότερα τίποτα δεν κάναμε πάλι. Ευχαριστούμε. Γιώργ. Ευχαριστώ. Ως εισηγήτρια Πρέπει να σας πω ότι φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την πρόταση που βασίζεται σε αυτή την ανθρωπιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Λοιπόν, για, τα διάφορες, για τους διάφορους ε, τομείς, επειδή πρόκειται για θέματα εσωτερική, ε, πρόκειται για εσωτερικές υποθέσεις, ε, έχουμε ήδη πει ότι φυσικά Είμαστε οι υπέρμαχοι αυτής της ανθρωπιστικής προσέγγισης για τους πρόσφυγες και για τους μετανάστες, αλλά ε, διαπιστώνουμε το Συμβουλίο δεν ε, έχει τις ίδιες ακριβώς απόψεις και πρέπει να ξέρουμε ποιες φωνές θα είναι πιο ηχηρές μέσα στο Συμβούλιο, ποια φωνή θα επικρατήσει. Εμείς πάντως από πλευράς ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να υποστηρίξουμε απαρέγκλητα αυτή την ανθρωπιστική προσέγγιση ε, για τους μετανάστες και για τους πρόσφυγες, ε, κυρίως σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε το Συμβούλιο να ακολουθήσει την ίδια κατεύθυνση. Γιατί μέχρι τούδε είναι πολύ διαφορετικά αυτά τα πράγματα που ακούμε από το Συμβούλιο και θα πρέπει να αλλάξει η προσέγγιση μας εν ώψη των διαπραγματεύσεων πώς θα καταπολεμήσουμε τους διακινήτες, πώς θα ενισχύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών και πώς θα συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή είναι ευκαιρία χρυσή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να θεωρούμε ως κάτι φυσιολογικό το φαινόμενο της μετανάστευσης. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Πρέπει να το διαχειριστούμε, ε, να αντιλήσουμε διδάγματα από το παρελθόν για να μην να αποφύγουμε το φαινόμενο, να το καλωσορίσουμε και να το διαχειριστούμε σωστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ο κ. Βασίρ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για την εξαίρετη παρουσίαση της κυρίας Κλάιν Σόλομον. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε δύο πράγματα, στους πρόσφυγες και στη μετανάστευση. Πρώτα, για τους πρόσφυγες. Ε, δουλεύουμε πάνω στο φάκελο που έχει να κάνει με τους απάτριδες Πήγα στον Μπαγκλαντές πριν από λίγο καιρό και είδα πάρα πολλούς πρόσφυγες που θέλησαν να βρούνε κάποιο καταφύγιο εκεί. Υπάρχουν 68 εκατομμύρια ε, πραγματικοί πρόσφυγες στον κόσμο και οι περισσότεροι από αυτούς ζουν στην χώρα που γεννήθηκαν ή στις γείτονες χώρες. Ένα εκατομμύριο ήρθε στην Ευρώπη πριν από μερικά χρόνια, αλλά 67 εκατομμύρια εξακολουθούν να ζουν στις χώρες που γεννήθηκαν ή στις γειτονικές, όπως η Ορδανία, το Λίβα, ο Λίβανος, η Τουρκία, το ο λιβανος η τουρκια το πακισταν και το Μπαγκλαντές. Οι χώρες ε, αυτές επομίζονται τεράστιο βάρος για να προσφέρουν εκπαίδευση σε αυτούς τους ε, ανθρώπους οι οποίοι θα τους μείνουν, γιατί δεν πρόκειται να επιστρέψουν στις χώρες τους, θα μείνουν πρόσφυγες σε αυτές τις γείτονε χώρες και κινδυνεύουν να γίνουν θύματα εκμετάλλευσης, γι' αυτό και χρειάζονται εκπαίδευση, χρειάζονται και δουλειές, στέγαση, ένταξη. Εμείς λοιπόν που είμαστε το πιο ανεπτυγμένο τμήμα του κόσμου πρέπει να βοηθήσουμε. Τώρα για την μετανάστευση τονίζω ότι ήρθε ο πατέρας μου στο Ηνωμένο Βασίλειο όχι ως πρόσφυγας, αλλά σαν οικονομικός μετανάστης. Έκανε έξι παιδιά. Και τα έξι έχουν τις δικές τους επιχειρήσεις ή τέλος πάντων πήραν σοβαρή εκπαίδευση και συνεισφέρουν τα μάλα στην βρετανική οικονομία. Πληρώνοντας φόρους βέβαια. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις επιτυχίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι που μετανάστευσαν. Τσαφέ, που είναι υφυπουργό στην κυβέρνησή μας, για παράδειγμα, έχει μια αντίστοιχη ιστορία. Ο δήμαρχος, και ολοκληρώνω πολύ σύντομα πρόεδρε, έλεγα λοιπόν ότι ο ίδιος ο δήμαρχος του Λονδίνου, ο Σαντί Καν, είναι επίση από τη μετανάστευση. Οπότε θέλω να πω, έχετε δίκιο. Η διαχείριση της μετανάστευση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι μετανάστες έχουν πολλά να προσφέρουν και πολύ σωστά μιλάτε για τις δημογραφικές ανάγκες των χωρών μας. Και γι' αυτό πρέπει να δεχτούμε τη μετανάστευση. Η μετανάστευση είναι επίση πάρα πολύ σημαντική λοιπόν. Ευχαριστούμε, Birgit Σίπελ. Η κυρία Σέπελ τα λέει με την κυρία Σαρτζεντίνη. Λόπες Αγγιλάρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Κλάιν Σόλομον για την παρουσίασή σας. Πρέπει να ξέρετε ότι πολλοί από εμά εδώ γνωρίζουν αυτά που γνωρίζετε, αυτά που μας λέτε, ότι η μετανάστευση δεν είναι κρίση, είναι μια ανθρώπινη διάσταση, πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Και ήρθε ο καιρός, οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν επικυρώσει τη συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία ρητά αναφέρεται στη διαχείριση της μετανάστευσης και θεωρείται είναι θέμα πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνομοθέτη για θέματα ασύλου, μετανάστευσης κλπ, αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης. Γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουμε τώρα την ευκαιρία όχι μόνο να δώσουμε νόημα στη διαχείριση της μετανάστευσης, χωρίς ε, να ενισχύουμε αυτό το ένστικτο κατά της μετανάστευσης, τα τελευταία δέκα χρόνια που ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας, δυστυχώς αυτό ακριβώ όμως γίνεται. Ο, τα κράτη-μέλη την αρνούνται, παρόλο που την επικύρωσαν. Αυτό ήθελα να πω λοιπόν. Εσείς είπατε πόσο σημαντικό είναι να δώσουμε μια ευκαιρία στην νόμιμη μετανάστευση, ιδίω αυτούς που για λόγους ανθρωπιστικούς ή άλλους τη χρειάζονται όχι μόνο αυτούς που θέλουν άσυλο ή τους πρόσφυγες, αλλά για ανθρωπιστικούς λόγους να ανοίξουμε τις πόρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν δεν υπάρξει αυτή η νόμιμη διαδρομή, δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν. Θα έρθουν, αλλά θα έρθουν διακινδυνεύοντας τις ζωές τους, των οικογενειών τους. Αγωνιζόμαστε σκληρά. Εγώ είμαι εισηγητής Προσπαθήσαμε πραγματικά σκληρά να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με το άρθρο 25 που, δημιουργεί, που προσφέρει τη δυνατότητα για εισόδους περιορισμένης διάρκειας για ανθρωπιστικούς λόγους. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να πετύχουμε και την ανθρωπιστική θεώρηση, τη βίζα. Με χώρες μέλη το μπλοκάρουν αυτό. Πρέπει να πιστούν και να καταλάβουν επιτέλους ότι πρέπει να βρουν ένα νόμιμο δρόμο, να τον φτιάξουν, μια νόμιμη διαδρομή για τη μετανάστευση. Αλλιώς αυτή τη συζήτηση θα την έχουμε και θα την ξαναέχουμε και δεν θα καταλαβαίνουμε τις πραγματικές συνέπειες της μετανάστευσης. Ευχαριστούμε, είπατε ξεκάθαρα τι εννοείται για την ανθρωπιστική βίζα. Λέω ο πρόεδρος, η Άννα Γκόμε έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ, Άννα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κλάιν Σόλομον. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο Μετανάστευσης να έχει να κάνει με τον πολιτικά ορθό λόγο, αλλά να κρύβει μια φοβερή πραγματικότητα, λέτε, να αντιμετωπιστούν οι αιτίε. Ωραία, είχαμε τους Νιγηριανούς εδώ, τις προάλλες, που είπανε με την Boko Χαράμ, με αποτέλεσμα πολύ να φεύγουν από τα σπίτια τους, ότι η πραγματική αιτία είναι τα όπλα και όχι αυτά τα οποία έχουν ξεφύγει από τη Λιβύα του Καντάφη, αλλά άλλα νέα ε, όπλα, ε, αυτοκίνητα με οπλισμό, τα οποία λένε ότι αγοράζουν και από την Ευρώπη. Αιθιοπία. Μια χώρα την οποία στηρίζουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί φορολογούμενοι με τα χρήματά τους. Και εκεί υπάρχει ένα καθεστώς που προχωράει σε φοβερή καταστολή. Και ελπίζω ότι αυτό το καθεστώς του θα πέσει σύντομα, γιατί γίνονται διαμαρτυρίες στους δρόμους ήδη. Εμείς με τα δικά μας τα χρήματα όμως πληρώνουμε αυτή την καταστολή, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή τους πάρα πολλοί νέοι στην Αιθιοπία. Θα μπορούσα να μιλήσω για τον Ήγερα που είχαμε μια αποστολή πρόσφατα. Αυτά που γίνονται εκεί δεν φτάνουν για να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα της νεολαίας να βρει ένα σκοπό στη ζωή της. Λιδί. Μα κορεδευόμαστε. Πληρώνουμε τους παραστευτικούς στη Λιβύη. Εσείς που έχετε κάνει εξαιρετικό έργο εκεί, που ο ΙΕ βρίσκεται εκεί, πόσοι ασχολούνται με την υπόθεση αυτή στη Λιβύη σήμερα από εσά. Τελικά καταφέρετε να διαχειριστείτε τους καταβλισμούς. Προφανώς όχι, εκεί γίνονται βασανιστήρια. Ε, προσπαθείτε που και που να σώσετε κανέναν αν μπορείτε. Οπότε κορυδεύουμε τους αυτούς μας και δεν είναι ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευση να μας πει την αλήθεια και να πάει στι κυβερνήσει μας και να την πει ομά. Πρόεδρος. Σίσιλ Κέγκε, ε, κύριε Σίπα, όχι δεν θέλει, εντάξει. Κύριε Σίπελ, καλά. Τη έκοψα τη φόρα. Σε εσύ λοιπόν που είναι συνεισηγήτρια με την κυρία Μετσολέ για τη μετανάστευση. Κανείς άλλος από την ΤΕΒΕ, ΑΦΕΤ που δεν έχει μιλήσει. Και μετά θα ακούσουμε και τη Λίντα που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης και φυσικά θα απαντήσει και η κυρία Κλάιν Σόλομον. Λοιπόν, αν κανείς άλλος θέλει το λόγο, τώρα να το πει. Όχι. Ωραία. Σεσίλια λοιπόν είναι τελευταία μιλήτρια. Ευχαριστώ Κλοντ, ευχαριστώ και εγώ την κυρία Κλάιν Σολομών, όχι μόνο για την πολύ εύστοχη ανάλωση που μας έκανε, αλλά και γιατί έθεσε το Κοινοβούλιο στο επίκεντρο της όλης διαδικασίας. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου ε, είναι πολύ σημαντικός κατά την άποψή μου σε όλες τις διαδικασίες, ε, όπως θα είναι πολύ σημαντικός και στην επόμενη ανανέωση των συμφωνιών της Κοτονού. Ε, ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Αλλά ε, τον θέσατε και στο επίκεντρο όσον αφορά τις επόμενες προκλήσεις μετανάστευσης. Πραγματικά εκτίμησα ιδιαίτερα την ολιστική σας προσέγγιση και όπως είπε και ο πρόεδρος μας ο Κλοντ, εμείς ε, προωθήσαμε ένα ψήφισμα για την ολιστική προσέγγιση στο Κοινοβούλιο, θέτοντας στο επίκεντρο, όπως είπατε και εσείς στην παρουσίασή σας, πολλά από αυτά τα σημεία. Ε, ευρύτατα θεματολόγια, ξεκινώντας από την έρευνα και τη διάσωση, τους νόμιμους διάβλους, ε, καταπολέμηση της ε, λαθροδιακίνησης ανθρώπων, ε, τις χώρες καταγωγής ε, μεταναστών και συνεργασία μεταξύ τους, ε, όλα τα θέματα ασύλου, για να φτάσουμε τελικά σε όλες τις πολιτικές και μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική ένταξη. Το γεγονός ότι τα θέματα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνίας μας σημαίνει ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού. Και είναι και κάτι το οποίο εκτίμησα ιδιαίτερα, μάλλον δεν άκουσα από την παρουσίασή σας, όρος κρίση. Αυτό σημαίνει ότι συνειδητοποίησαμε ότι δεν θα πρέπει να έχει χώρο εδώ, διότι εμείς πρέπει να τοποθετήσουμε τη συζήτησή μας σε ένα όραμα το οποίο αφορά μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ε, ε, προτάσεις. Φυσικά υπάρχει και μια επίγουσα ανάγκη ε, την οποία πρέπει να λύσουμε ταχύτητα. Έχω τις δύο, εξής δύο ερωτήσεις. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ιδέα των κλιματικών προσφύγων με την βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών. Δεν αναφέρομαι στα όσα ανέφεραν οι συνάδελφοι. Πώς μπορούμε να φτάσουμε όμως σε αυτή την ορολογία, τη χρήση του όρου των κλιματικών προσφύγων. Και δεύτερον, ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αφρικανικής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία παγκόσμια ε, συμφωνία και επομένως οι δύο αυτοί οι παράγοντες δεν μπορούν να μην συμμετέχουν. Οι πολιτικές μας ε, για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες ή τους ανθρώπους που ζητούν ε, διεθνή προστασία πρέπει να είναι ίδια. Και ολοκληρώνω λέω ότι, λέγοντας ότι θα πρέπει να έχουμε και να αντιτάξουμε κάποια επιχειρήματα σε όλο αυτό το αφήγημα πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Εχθές αποφασίστηκε ότι ως ομάδα σοσιαλιστών και δημοκρατών θα προτείνουμε ένα ψήφισμα για το ε, Παγκόσμιο Σύμφωνο Μετανάστευσης ε, και το Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες ε, και νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Κλάιν Σόλομον για να απαντήσει. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Ε, έχετε 6-7 λεπτά λοιπόν για να απαντήσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ όλους για το πάθος ε, με το οποίο τοποθετηθήκατε. Ε, ήταν εύλογα τα σχόλιά σας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε μεταξύ άλλων και η κυρία Γκόμες. Νομίζω ότι σε σχέση με αυτήν την κρίση που σχετίζεται με τη μετανάστευση και κυρίως με τους πρόσφυγες, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι φυσικά ότι το βασικό είναι να καταπολεμήσουμε τις αιτίες. Ε, το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση φυσικά δεν θα πρέπει να καλύψει τις, τις πραγματικές αιτίες για τις οποίες φεύγουν από τη χώρα τους ε, οι άνθρωποι, γιατί πέρα από τη Σύμβαση για τους πρόσφυγες, ακόμη και γενικότερα ως προς τη μετανάστευση, υπάρχουν τα θέματα βίας, ε, διαφορά και αυτές είναι οι βασικές αιτίες μετακίνησης αλλά και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οι κλιματικές αλλαγές. Αυτά τα θέματα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μόνο στη ρίζα τους, καταπολεμώντας τη ρίζα αυτών των αιτιών και γι' αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο δεν θα πρέπει να ε, καλύψει αυτές τις ε, ευθύνε ε, για τον κρατών μελών και για τη διεθνή κοινότητα που πρέπει να υπομισθούν την ευθύνη να μειώσουν αυτή την πίεση διότι δεν έχουν την επιλογή, είναι απεγνωσμένοι και προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτές τις καταστάσεις. Γι' αυτό μετακινούνται οι άνθρωποι. Ε, επίσης, όλο είναι και περισσότερο να γνωρίζουμε ότι αυτοί που καταναγκαστικά αποχωρούν από τη χώρα τους ε, ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό εντοπίζονται το εσωτερικά στη χώρα τους για κλιματικούς λόγους, λόγους κλιματικών αλλαγών. Αλλά τώρα δεν είμαι σίγουρη ότι θα ήταν καλό να φτιάξουμε νέα κατηγορία ε, τέτοιων ε, μεταναστών. Μην ξεχνάμε όμως ότι πολλοί δεν μπορούν είτε προσωρινά είτε μόνιμα να επιστρέψουν ε, στη χώρα προέλευσης λόγω υποβάθμισης του περιβάλλοντος και λόγω κλιματικών αλλαγών. Και άρα θα πρέπει να προβλέψουμε ε, μεγαλύτερη προστασία. Αυτή τη στιγμή προσφέρεται προσωρινή προστασία και σίγουρα με πιο συστηματικό τρόπο θα μπορούσαμε να έχουμε εναρμονισμένα κριτήρια για τέτοιου είδους μέτρα προστασίας ε, για κλιματικούς λόγους και πιστεύω ότι ε, το παρόν φόρουμ, το Κοινοβούλιο και οι Επιτροπές σας μπορούν να ε, συμβάλλουν τόσο ώστε αυτοί που δεν έχουν επιλογή και αναγκάζονται να διαφύγουν να τύχουν προστασίας για τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης και το βάρος που έχουν στη δημόσια συζήτηση. Κυρία Μούντι. Σας ευχαριστώ διότι υπογραμμίσατε αυτό που ουσιαστικά είναι ευνόητο όταν βλέπουμε τις προβολές για το μέλλον. Ε, οι νέοι θα πρέπει να συμβάλλουν ε, φυσικά στις, στα συνταξιδοτικά συστήματα για να διασφαλίσουν την βιωσιμότητά τους. Αυτό φυσικά είναι ε, καταφανές και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη και αν υπάρχει αυξημένη κινητικότητα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν το μήνυμα θα πρέπει να περάσει ε, στο κοινό. Ε, και αυτό σχετίζεται επίσης με αυτά που είπατε πολύ, δηλαδή με ποιο τρόπο μπορούμε με πιο λογικό τρόπο να βασιστούμε σε συγκεκριμένα αυτά στοιχεία για να συνεχιστεί η δημόσια σε συζήτηση, διότι κυριαρχείται από συναισθήματα αυτή τη στιγμή, από τον φόβο, το φόβο για το αλότριο, ε, το φόβο για κάποιον που δεν μιλάει την ίδια γλώσσα, δεν έχει το ίδιο θρήσκευμα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ε, ειλικρινείς. Υπάρχει ε, η Ισλαμοφοβία και ραντισμό σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στη... Χαρακτηρίζεται αυτό τη δημόσια σκηνή και φυσικά είναι μια κλίση ε, ανθρώπινη φυσική. Δηλαδή φοβούμαστε το αλότριο. Ναι, αλλά ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος ε, των εθνόντων των πολιτικών και κυρίως ε, των βουλευτών. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά τα βασικά ανθρώπινα ένστικτα, διότι μόλις περάσουμε αυτή την επιφάνεια, το, το επιφανειακό στρώμα, όλοι οι άνθρωποι είμαστε και ε, μπορούν οι μετανάστες με το επιχειρηματικό τους πνεύμα, με την προσήλωσή τους στην κοινωνία υποδοχής να συμβάλλουν ε, στα ε, κοινωνικά δρόμενα. Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας, ε, διότι πρέπει να αποδομήσουμε αυτό το φόβο, αυτή την ενστικτόδη ατυχή ομολογουμένως αντίδραση υπάρχουν ναι, αποδεικτικά στοιχεία με ε, έκθεση, πρόσφατη έκθεση McKinsey, επίσης από το Intelligence Unit του Economist, μια άλλη εξαρτική έκθεση όπου βλέπουμε συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία. Δυστυχώς όμως ε, το κοινό δεν αντιδρά σε αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει αυτή η συναισθηματική διάσταση που κυριαρχεί και μην ξεχνάμε ότι ε, προεκλογών οξύνονται τα πνεύματα και γι' αυτό ε, ηγετικός ρόλος, πολιτικός ρόλος ε, ε, χρειάζεται για τους βουλευτές ούτως ώστε να αποδομηθούν αυτοί οι μύθοι ε, και ανεξαρτήτως θρησκεύματος και ε, φιλετικής προέλευσης να συνειδητοποιήσουμε ότι μιλάμε για ανθρώπους που μπορούν με καινοτόμο τρόπο να συμβάλλουν διότι έχουν ικανότητε ε, και η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών, αυτοί που μετακινούνται, ε, συνήθως είναι αυτοί που, έχουν, που είναι και πιο ανθεκτικοί, που ε, αναλαμβάνουν κάποιο κίνδυνο για να πετύχουν κάτι. Δηλαδή το είδο των ανθρώπων που θα θέλουμε να βλέπουμε σε ευρωπαϊκέ κοινωνίε ε, που θα δημιουργήσουν νέε επιχειρήσει, θα δημιουργήσουν θέσει εργασία, θα βρουν στα προβλήματα. Αυτή είναι η πηγή τη καινοτομία, λοιπόν, σε πάρα πολλές χώρες και γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτό τον ηγετικό ρόλο. Εμείς να σα δώσουμε τα στοιχεία, τη βάση ε, των απτών στοιχείων, αριθμητικών στοιχείων, όμως σε πιο συναισθηματικό επίπεδο πρέπει να επιδιώξουμε μία αντίδραση και πρέπει να ξεπεράσουμε τη φιλετική προέλευση και το θρήσκευμα και τα ε, πιστεύω του καθενό, διότι δεν είναι αυτέ απειλέ για, ε, για το κράτο δικαίου, για τις αρχές που εγγράφονται στα συντάγματα και στις ένομες τάξεις για την ε, κατάργηση των διακρίσεων και αυτό συνδυάζεται φυσικά με τις δίκαιες κοινωνίες και το στόχο για την κατάργηση των αποκλεισμών. Και τέλος, ε, για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση. Ξέρουμε πως ε, ως προς την εκπόνηση πολιτικών. Πολλοί ε, συντονίζονται με τις προεκλογικές καμπάνιες και αυτό συμβαίνει ακριβώς τώρα. Λοιπόν, από πλευράς οικονομικής, όταν πάσχουμε από ανεργία, δύσκολα κάποιος να ισχυριστεί ότι η λύση είναι να ε, επιδιώξουμε περισσότερους νόμους διάβλους. Όμως ε, όλα αυτά είναι χρονοβόρα και θα πρέπει ήδη τώρα να δράσουμε για να προβλέποντας για το μέλλον και θα πρέπει με ρεαλιστικό τρόπο να κάνουμε μια αποτίμηση για το μέλλον. Πού θα υπάρχουν τα χάσματα, τα κενά Ω προ τι δεξιότητε, ε, όταν μιλάμε για υψηλέ δεξιότητε, στον τομέα τη πληροφορική παραδείγματο χάρη. Και όχι μόνο και σε, σε χαμηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων, διότι η πραγματικότητα πια είναι σε πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες και σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες οι υπήκοοι δεν ενδιαφέρονται πλέον, δεν ε, θέλουν να εργάζονται σε αυτούς τους ε, τομείς, σε χαμηλών δεξιοτήτων, στον τομέα της υγείας, σε περίθαλψη των παιδιών, ε, στην εστίαση, ε, στη γεωργία. θα χρειαστούν λοιπόν περισσότεροι άνθρωποι σε αυτούς τους τομείς, χρειάζεται αυτές τις δεξιότητες και το εργατικό δυναμικό και στα δύο επίπεδα, σε χαμηλό και σε υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων. Και αυτό όμως πρέπει να το προγραμματίσουμε εκ των προτέρων. Και μπορούμε να διαχειριστούμε, και αυτό το λέω από πρακτική σκοπιά και πολιτική πλευρά, Χρειάζεται προγραμματισμός και συνεργασία κυρίως με τις χώρες προέλευσης, ούτως ώστε να προετοιμάσουμε τις μετανάστες για αυτή τη νέα εμπειρία, για να έχουν τις διεξιότητες και τις πολιτιστικές δυνατότητες να γνωρίζουν όχι μόνο τα δικαιώματα, αλλά και τις ευθύνε που θα έχουν όταν έρθουν. Η βιομηχανική κλάδη, τα κράτη μπορούν να συνεργαστούν σε αυτό το επίπεδο, ούτως ώστε όσοι έχουν τις αποτελούμενες δεξιότητες, όσοι θέλουν να βρουν να σε κάποια χώρα να βρουν κάποιον από την οικογένειά τους με την επανένωση να είναι προετοιμασμένοι. Έτσι μπορούμε να αποφύγουμε την εκμετάλλευση, την βία, διότι πότε υπάρχει εκμετάλλευση, όχι μόνο με τους ε, λαθροδιακινητές. Μην το ξεχνάμε, αλλά και με αυτούς που προσλαμβάνουν ε, τους μετανάστες ε, και τους εκμεταλλεύονται κατάφορα με υψηλότητα μισθόδοντα, επίσης ε, όσοι τους απασχολούν παράνομα και δεν τους επιτρέπουν έτσι να προστατεύονται από την εθνική εργατική νομοθεσία. Υπάρχει λοιπόν μια ε, μεγάλη σύγκληση συμφερόντων για την σωστά ρυθμισμένη μεταναστευτική ροή προ όφελο ε, και των ατόμων και των κοινωνιών. Για την ανθρωπιστική διάσταση, το 2015 με λύπη διαπιστώσαμε, όπως είπατε και εσείς κύριε Μπαζίρε, ένα πολύ ε, μικρό αριθμό σε σχέση με το παγκόσμιο αριθμό ε, ε, προσφύγων να έρχονται στην Ευρώπη. Μα ήταν προβλέψιμο αυτό. Αν δείτε ποιε συνθήκε ίσχυαν στην Τουρκία, στην Ιορδανία, στο Λίβανο, δεν είχαν καμία άλλη προοπτική. Αν του είχαμε δώσει τότε νόμιμος διάβιου για τη μετανάστευση, θα είχαμε σώσει πάρα πολλέ ζωέ και φυσικά όλα αυτά τα προβλήματα που προέκυψαν. Αυτά τα πραγματικά πράγματα μπορούμε να τα προβλέπουμε, να τα διαχειριζόμαστε, να τα προγραμματίζουμε και να τα διαχειριζόμαστε με τρόπο εποφελές, συγγνώμη, για τα άτομα αυτά και για τις κοινωνίες. Δηλαδή χρειαζόμαστε καλύτερα εξορροπημένες πολιτικές δομές. Όχι αυτή την αρνητική ε, αντίδραση που διακατέχεται από ρατσισμό και από <clears throat>